El señor presidente. Επαναλαμβάνεται η αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχά Καταρχάς, έχω να σας ανακοινώσω ότι έχουν διανεμηθεί τα χθεσινά συνοπτικά πρακτικά και αν δεν έχετε παρατηρήσεις ε, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Προχωρούμε. Έκθεση Κοέγιο χαρακτηριστικά ασφαλείας και χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Το λόγο έχει ο εισηγητής, κύριος Κοέγιο. Για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ.